Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Ελπίζω να είσαστε όλοι έτοιμοι και να έχετε και καλές διακοπές και με ενθουσιασμό να έχετε επιστρέψει για δουλειά εδώ. Το πρώτο θέμα που έχουμε είναι την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τότε εγκρίνεται χωρίς τροποποίησης. Δεν βλέπω εδώ καμία αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν. Επόμενο θέμα. Ανακοινώσεις. Η προθεσμία για τροπολογίες για τον κανονισμό όσον αφορά διάφορες νομικές πράξεις για τις ρυθμιστικέ διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το άρθρο 290 και 291 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τροπολογίες έχουν κυκλοφορήσει από τον εισηγητή στην ΕΒΗ χτε, 30 Αυγούστου. Και όπω έχουν ζητήσει κάποιε ομάδε η προθεσμία ανοίγει για τροπολογίε. Θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή μας, ΕΝΒΗ, και ίσως και επιστολή από τον πρόεδρο της ΕΝΒΗ προς την Νομική Επιτροπή. Το χρονοδιάγραμμα θα έχει ως εξής. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στην Επιτροπή μας ΕΝΒΗ είναι η 6η Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα. Ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ θα λάβει χώρα την 28η Σεπτεμβρίου και η προθεσμία για τροπολογίες στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Άλλη ανακοίνωση. Ακύρωση της συνεδρίασή μας το απόγευμα της 7 η Σεπτεμβρίου. το σχέδιο τη ημερήσια διάταξη για το πρωινό τη 7η Σεπτεμβρίου. Θα σα τελείωσω γιατί πιο γρήγορα. Τώρα, αλλαγέ στη γραμματεία τη ΕΝΒΗ. Ο γιο Φερφλούτ, ο οποίο δούλευε στη γραμματεία τη ΕΝΒΗ για πάνω από 10 χρόνια, συνταξιοδοτείται από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά από πάνω από 40 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκ μέρους λοιπόν της Επιτροπής μας θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το έργο του εδώ και για τη στήριξή του στο έργο μας όλα αυτά τα χρόνια. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Διερμηνία. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες. Με εξαίρεση τα στονικά, τα λετονικά, τα μαλτέζικα και τα γκέλικ. Ως συνήθως τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και επίσης η συνεδρίασή μας μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Επόμενο. Συστάσεις συντονιστών της 7ης Ιουλίου έχουν κυκλοφορήσει οι συστάσεις αυτές ηλεκτρονικά. Οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού, υποκατάστατα του συνόλου του διατολογίου. Η Τζούλι Γκέρλινγκ και η Άννη Σχρέιερ Πίρικ είναι οι συνεισηγήτριες. Θα δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στην κυρία Γκέρλινγκ. Παρακαλώ κυρία Γκέρλινγκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. παρακολούθησα το θέμα αυτό και στα πλαίσια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου υπό την επιμέλεια και την εισήγηση της κυρίας Ρης. Είχαμε λοιπόν ζητήσει το θέμα και στο παρελθόν. Έμειναν κάποια θέματα σε εκκρεμότητα και τα θέματα αυτά δημιουργούνται γιατί κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικούς προσανατολισμούς, παραδόσεις και τρόπους με τους οποίους έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι χαμηλές σε υδατάνθρακες διατροφές και δίαιτες στην Ευρώπη. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στην φάση όπου έχει προχωρήσει αρκετά το πράγμα. Ίσως για πολλούς να φαίνεται εξαιρετικά περίπλοκο και λαβυρινθώδες. Τέσσερα χρόνια το συζητάγαμε ουσιαστικά. και ίσως να αναφέρομαι σε κάποια θέματα τα οποία να μην παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά επανειλημμένα. Ε, μπορεί κανείς να υποστηρίξει, είναι η άποψή μου, αυτών των, ε, αυτές τις τροφές ε, Υποκατάσταση συνολικά της ε, διατροφής, των αναγκών διατροφής, γιατί βοηθούν αυτούς οι οποίοι είναι υπέρβαροι να χάσουν τα κιλά τα οποία ε, απαιτείται να χάσουν. ιδιαίτερα για τους πολίτες οι οποίες είναι σε προχωρημένα στάδια παχυσαρκίας και γι' αυτό λοιπόν τα προϊόντα αυτά έχουν αποδείξει ότι με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και χωρίς συνέπειες υγείας βοηθούν η αρχία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα όπως διαβήτη και δημιουργεί επιβαρύνσεις για τα συστήματα υγείας και γι' αυτό ακριβώς τέτοιου είδους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων πρέπει να τους υποδεχθούμε θετικά. Υπάρχουν υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας. Σε πολλές χώρες τα ποσοστά αυτά φτάνουν of national healthcare budgets in the EU. There's a very big chunk of health spending that if we were to uh, Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά παχής αρκείας και στη δική μου χώρα η υπέρβαρη είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χειρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χρησιμοποιείται και η μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω της υποκατάστασης όλων των διατροφικών αναγκών από συγκεκριμένα προϊόντα διατροφής. Υπάρχουν κάποια, θα έλεγα, κάποια, κάποιες συζητήσεις, όχι αποδεδειγμένες όμως και όχι τεκμηριωμένες, ότι τα προϊόντα αυτά δημιουργούν διατροφικές διαταραχές και οδηγούν πολλές φορές στην πλήρη απίσχναση των συγκεκριμένων προσώπων. Αλλά δεν είναι κάτι το τεκμηριωμένο. Δεν ε, η σύσταση αυτή λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο απορρίπτω, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται σωστή διαχείριση, προσεκτική διαχείριση, να δούμε τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η υποκατάσταση της συγκεκριμένης ρύθμισης Το θέμα δεν είναι ε, να δούμε πόσο εφικτές είναι οι προτάσεις αλλαγών που γίνονται από πλευράς των κατασκευαστών και ε, δεν είναι να πούμε εμείς ε, ποια θα είναι η μορφή, η υφή, η γεύση των προϊόντων υποκατάστασης. Πάντως Τα προϊόντα αυτά πρέπει να τηρούν ορισμένες παραμέτρους και πρέπει να σέβονται ορισμένα χαρακτηριστικά. Είπαμε, η εμφάνιση, η υφή και η γεύση δεν είναι αυτό το οποίο που μας ενδιαφέρουν. Η χρηστικότητα και το εφικτό της παραγωγής των προϊόντων αυτών μας ενδιαφέρει από πλευράς διατροφικών χαρακτηριστικών. Γίνονται λοιπόν συστάσεις για την αλλαγή στο περιεχόμενο των προγραμμάτων και υπάρχουν μερικές φορές αντιδράσεις από πλευράς των κατασκευαστών οι οποίοι θεωρούν ότι με τις αλλαγές αυτές τα προϊόντα τους δεν θα είναι πλέον ε, εμπορεύσιμα, δεν θα είναι φαγώσιμα ουσιαστικά και αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι ουσιαστικά τα προϊόντα αυτά να φύγουν από την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν στη συνολική πρόταση έχω την στάση αυτή η οποία είναι απορριπτική αλλά επαναλαμβάνω ότι για κάποια κριτήρια διαφωνώ και δεν διαφωνώ σε σχέση με κάποιες από τις προτάσεις αυτές για το περιεχόμενο των προϊόντων και δεν θα πρέπει οι αλλαγές αυτές, οι οποίες δυστυχώς έτσι όπως έχουν τώρα, καθιστούν το προϊόν μη ελκυστικό σε επίπεδο εμφάνισης και γεύσης, μειώνουν τη ζωή διάρκειας, την διάρκεια ζωής συγγνώμη, του συγκεκριμένου προϊόντος στα ράφια των καταστημάτων και τα καθιστούν, εν πάση περιπτώσει, μη βρόσιμα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι θέλουμε εμείς περισσότεροι υπέρβαροι ε, να ε, χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά ή θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια χαρακτηριστικά που θα μίκριναν τον αριθμό αυτό. συνήθως ακολουθούνται διατροφικά προγράμματα τα οποία πάρα πολύ σπάνια καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του προσώπου, του ασθενούς και οδηγούνται οι καταναλωτές σε υπερβολές. Φυσικά και οι υπερβολές αυτές θα πρέπει να αποφευθούν και εδώ ακριβώς τίθεται το θέμα των προϊόντων. Υπάρχει επίσης και το θέμα της πώληση στο διαδίκτυο των προϊόντων, σαφώς και θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να έχουμε προϊόντα τα οποία να είναι ελκυστικά λοιπόν για τους καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις εμπειρικές ε, ε, γνώσεις και ε, θα έλεγα και τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει και η σύσταση ως έχει τώρα είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει τους αρχικούς της στόχους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η κυρία Γκροσετέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τη στήριξή μου στα λόγια της κυρίας Κιάλη και θα ήθελα να εκφράσω και τις ανησυχίες των συνεισηγητών σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο για τις κατεξουσιοδότηση πράξης με, με τους ορισμούς των τριών κριτηρίων για την υποκατάστατα γευμάτων Έχω την εντύπωση ότι παραμελούμε και αφήνουμε κατά μέρο ορισμένες παραδοχές πολύ σοβαρές που ε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να είναι λιγότερο διαθέσιμα αυτά τα προϊόντα, αυτά τα υποκατάστατα γευμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για μεγάλο μέρος του ε, πληθυσμού που πάσχει από το να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο έχουμε αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν αυτά δίδονται χωρίς να ακολουθούνται οι συστάσεις και χωρίς να υπάρχει παρακολούθηση ιατρική. Τα υποκατάστατα γευμάτων αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται αυστηρά. Τα νέα κριτήρια για τη σύνθεση των υποκαταστάτων αυτών, όπως προτείνονται στο σχέδιο για την κατεξουσιοδότηση πράξη, κατά τη γνώμη μου μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στη γεύση και στην οσμή και στην ουσία τελικά αυτών των προϊόντων, και ουσιαστικά ε, με αυτές τις προϋποθέσεις το κόστος θα εκτοξευθεί. Δεν βλέπω πώς αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για τους υπέρπαρους ή τους παχύσαρκους να τα προτιμήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βασίσει τη δουλειά της στην ανάλυση της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η ίδια η υπηρεσία αναγνωρίζει ότι από τα ισχύοντα κριτήρια για το γενικό πληθυσμό έχει εικάσει ε, αντίστοιχες προβλέψεις για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Και αυτό αγείρει πολλά ερωτηματικά. Γι' αυτό και στηρίζω την πρόταση της κυρίας Γκέρλιν. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ η κυρία εσάντων Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι διότι το ΕΛΚΑ αναγνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ε, αρκείας στην Ευρώπη αλλά και ατόμων που είναι υπέρβαρα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται συζήτηση σε, ευρω... σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τι δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε για να καταπολεμήσουμε αυτή την επιδημία παχυσαρκίας να ασχοληθούμε με το θέμα, να συμφωνήσουμε κάτι να κάνουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το συγκεκριμένο φάκελο, τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η δική μας πολιτική ομάδα στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν στηρίζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν πράγματα, να αναλυφθούν δράσεις σε αυτό τον τομέα και αναφορικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απαραίτητες αντενδείξεις και να τίθενται σε εμπορία με τον πιο ορθό τρόπο, στο βαθμό του εφικτού. Ναι, να υποκαθιστά κανείς ένα από τα γεύματά του καταναλώνοντας αυτά τα προϊόντα. Να το πράττει όμως σε διάλογο και κατόπιν διαβούλευσης με τους επαγγελματίες της υγείας οι οποίοι και θα καθοδηγούν τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Ορισμένες τροπολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράγματι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την μυρωδιά, ε, την οσμή ή το γεύση που έχει κανείς όταν καταναλώνει αυτά τα προϊόντα. Όμω θα πρέπει να είναι σε θέση η παραγωγή να προσαρμοστούν στις νέες προϋποθέσεις. Όσο σοσιαλιστέ και δημοκράτες είμαστε πεπισμένοι ότι είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει τέτοια πρόταση, είναι καλό το ότι επιμένει ε, να υπάρξουν συστάσει και ενδείξεις για την θρεπτική ε, σύνθεση όλων αυτών των προϊόντων. Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και όσα ευχαριστώ η κυρία Πεντιτσίνη, παρακαλώ. Πεντιτσίνη. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Έχετε το λόγο. Και στη δική μου χώρα, στην Ιταλία, όταν κάποιος είναι παχύσαρκος, το θέμα των υποκατάστατων διατροφής είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεν χρησιμοποιούνται τα προϊόντα αυτά μόνο όμως για τους παχύσαρκους αλλά και για κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι ίσως να έχουν μια μικρή επιβάρυνση στον τομέα του βάρους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη σημερινή συζήτηση. Από τη μία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι λίγο θα έλεγα αφαίρετα ο καθορισμός των στόχων, ο καθορισμός των θεωρητικών μέσων που υιοθετούνται για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα αυτά, συμπεράσματα όμως τα οποία θα έχουν απτές, ε, απτά αποτελέσματα και επιπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν μιλάμε για τοξικά προϊόντα, για ουσίες τοξικές, αλλά για προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την βοήθεια ως προς την αποκατάσταση της υγείας ενός τμήματος του πληθυσμού. Είναι υπερβολικό λοιπόν να πούμε ότι τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να, ίσως να εμποδίσουν α, τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει επενδύσεις να συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα τους. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με την άποψη η οποία ακούστηκε ήδη για το θέμα της σύνθεσης των υποκαταστάτων γιατί οι νέες ρυθμίσεις θα περιορίσουν την διαθεσιμότητα των προϊόντων αυτών. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσουν να καθορίσουν με διαφορετικό τρόπο τα ανώτατα ποσοστά περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, άλατα και ε, λίπη. Τώρα, σχετικά με την απαγόρευση α, ε, χρήσης των προειδοποιήσεων για θέματα υγείας, γιατί υποτίθεται ότι η κατάσταση στην ετικέτα όταν είναι αναλυτική επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές οι οποίες χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε πλήρως αυτό, αυτή την πρόταση. Η κυρία Ρίση έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Είμαι εισηγήτρια από πλευράς ε, των φιλελεύθερων και ήμουνα και πριν από τέσσερα χρόνια, όπως το υπενθύμησε και η κυρία Γκέρλινγκ, για όλα αυτά τα υποκατάστατα, για αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία πληθυσμού. Φυσικά και συμμερίζομαι την επιθυμία όλων μας να καταπολεμήσουμε την μάστιγα αυτή της παχυσαρκίας, όμως αναρωτιέμαι για τον τρόπο που έχει προτιμηθεί από τις συνεισηγήτριες, την κυρία Γκέλ και την κυρία Σχράιερ. Τι κάνει με την κατεξοδότηση πράξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστέρησε τόσο πολύ. Είχε λόγους βέβαια που το καθυστέρησε. Έγιναν συζητήσεις με τους διάφορους κλάδους. Τι κάνει λοιπόν η Επιτροπή. Θέτει ε, κάποια όρια βάσει των πληροφοριών που έχει πάρει, όπως είπε και η κυρία Γκέρλινγκ, για τον τρόπο με τον οποίο ε, παράγονται τα προϊόντα αυτή αναφέρονται διάφορα πλονεκτήματα στο κείμενο, καλύπτουν όχι μόνο τις ε, δίαιτες ε, με χαμηλές θερμίδες, αλλά και άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και τις περιπτώσεις ε, των διαιτών που είναι κάτω από τις χίλιες θερμίδες. Και το είπανε πολύ μέχρι τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια καινοτομία ότι απαγορεύει ισχυρισμού ότι κάνουν τα προϊόντα αυτά καλό στην υγεία. Αυτό είναι το καινούργιο και είναι πολύ αυστηρή η Επιτροπή συνολικά για τους ισχυρισμού των διαφόρων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λοιπόν τα προϊόντα αυτά χωρίς συνταγή από γιατρό, μέχρι 8 εβδομάδες το πολύ. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να ξέρουμε ότι η εμπορία των προϊόντων αυτών και η πώλησή τους δεν πρέπει να γίνεται έτσι άκρατα σε πολίτες οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι. Τώρα άκουσα τα επιχειρήματα για την αντίρρηση, έτσι. Άκουσα τα επιχειρήματα, ναι, είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό και που ίσως να είναι προβληματικό. Όλοι οι πυρογνώμονες, εδώ δώσαμε την εντύπωση ότι όλοι λίγο πολύ δεν συμφωνούν. Μα δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Γιατί άκουσα και εγώ πολλούς που λένε ότι η βιομηχανία φτάνει να, όπου να να παρουσιάσει στην αγορά προϊόντα τα οποία να έχουν την γεύση την επιθυμητή. Το άλλο θέμα είναι το κόστος βέβαια. Οι αλλαγές που προβλέπονται θα έχουν επιπτώσεις στο κόστος, οι πρωτενικές αλλαγές για παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θα ρυθμιστεί από την ίδια τη βιομηχανία και μια μικρή αύξηση 5 σαντίμ για παράδειγμα για τα προϊόντα αυτά είναι ένα ποσό που μπορεί να διαθέσει το κοινό το οποίο ενδιαφέρεται Συνεπώς, πιστεύω ότι νομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δούλεψε σωστά. Είχε βέβαια μέχρι τον Ιούλιο του 2015 για να προχωρήσει στους κανόνες αυτούς σύνθεσης και ενημέρωσης. Αν καθυστέρησε, είναι εξαιτία της συζήτηση με την βιομηχανία και τον κλάδο που ήταν πολύ επιφυλακτική να δεχτεί την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας Τροφίμων. Είναι πράγματι βλέπουμε ότι ο κλάδος επιμένει στις θέσεις του. Πέντε χρόνια είχαμε προβλέψει στον τριμερή διάλογο. Δεν ήταν κακό για την προσαρμογή. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι φτάνουμε στο 2022 και ο κλάδος λέει ότι δεν φτάνει. Εδώ νομίζω το παρακάνουμε. Τέλος. Εδώ έχουμε μπροστά μας μια γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων που την παρακολούθησαν και οι εμπειρογνώμονες 27 χωρών μελών. Έτσι, γιατί δεν υπόθηκε αυτό μέχρι τώρα. Τα προβλήματα, από ό,τι φαίνεται, προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Αυτό πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, οπότε προτείνω μια που ήμουνα και παλιά εισηγήτρια για τέτοια προϊόντα, προτείνω να μην στηρίξουμε την αντίρρηση και να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιθυμία της να συνεχίσει το έργο το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 2013 με την πρώτη κύρια νομοθεσία και με την συνέχεια που δόθηκε και έχουμε φτάσει εδώ στην κατεξοδότηση αυτή η πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έικιν ο Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να χαιρετήσουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα της παχυσαρκίας. Τώρα το κατά πόσο η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα στεφτεί από επιτυχία ή όχι, αυτό με είναι αποδειχτή. Η κατάσταση δίχως άλλο είναι αρκετά επίμαχη. Γιατί τελικά ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία εκτός από τη ζάχαρη, τους υδατάνθρακες, μας επιτρέπουν να χάσουμε βάρος. Πρόκειται για ζωικά τρόφιμα βασικά και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ θα έπρεπε να ξαναδεί την πρότασή της γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της επαρκώς αυτή την πτυχή. Ότι δηλαδή τα προϊόντα που κάνουν ε, τον κόσμο να παχαίνει βρίσκονται ελεύθερα στην αγορά και συχνά τα φρούτα και τα λαχανικά κοστίζουν πιο ακριβά από το κρέας, το γάλα και άλλα. Συνεπώς, ο κόσμος τελικά αναγκάζεται να περιοριστεί, να καταλήξει, να τρέφεται με τυριά, φτηνά τυριά ή με φτηνό κρέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου λοιπόν, να ασχοληθεί με αυτά τα προϊόντα θα έπρεπε να φροντίσει αυτά να είναι πιο ακριβά και να μειώσει τις επιδοτήσεις της γεωργικές για αυτού του είδους τα προϊόντα. Τότε ίσως φτάναμε πιο εύκολα σε λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να εξετάσει αυτή την κατάσταση. Πιστεύω επίσης ότι θα έπρεπε να στραφεί όλο και περισσότερο στην ε, ε, πρόθεση των, ε, της χορτοφαγίας και της χορτοφαγίας χωρίς ε, καθόλου κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Να αλλάξουμε συνήθειες ζωής, διατροφής. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση δηλαδή, αυτή που σας εξήγησα στην αρχή. Ότι από τη μια λέμε ότι θέλουμε μια πιο απόλυτη προσέγγιση για να αλλάξουμε τις ε, τροφικές ε, συνήθειες των επόμενων γενιών, αλλά αυτό θα γίνει μόνο εάν εγκαταλείψουμε τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στραφούμε σε φυτικά προϊόντα και μόνο τα οποία παράγονται με οικολογικό και βιολογικό τρόπο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό στο οποίο καταλήγουμε εδώ είναι ότι χρειάζεται πιο σαφής ε, ρύθμιση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα υποκατάστατα. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά πρέπει να ξέρουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται και να συνενούν στη χρήση τους. Εδώ μιλάμε για την παχυσαρκία και τους υπέρβαρους. Σε πολλές χώρες τέτοια προϊόντα χρησιμοποιούνται και από άλλους ανθρώπους, όχι μόνο από παχύσαρκους και υπέρβαρους, οπότε καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου τα προϊόντα αυτά είναι εύκολα προσβάσιμα από οποιονδήποτε και με ισχυρισμούς οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικοί και τελικά μπορεί να εξαπατούν τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος τι υπάρχει μέσα στο προϊόν που αγοράζουν, ποιες είναι οι πρωτενικές ε, και άλλες ε, ουσίες που περιλαμβάνουν και θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε την αντίδραση σε διάφορα πράγματα που ακούσαμε. Δηλαδή, θα καταλήξει η πρόταση της Επιτροπής σε μικρότερη προσφορά τέτοιων προϊόντων προς τους καταναλωτές. Θα καταλήξει σε υψηλότερο κόστος. Ε, θα οδηγηθούν ε, οι καταναλωτές σε άλλα προϊόντα περισσότερο επικίνδυνα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που τέθηκαν εδώ. Καλό θα ήταν η Επιτροπή να μας τα απαντήσει και να δούμε έτσι ποιε θα είναι οι συνέπειες για τους καταναλωτές και κατά πόσο θα μειωθεί η δυνατότητα των καταναλωτών να καταπολεμήσουν ε, την παχυσαρχία τους. Καλό θα ήταν να έχουμε λοιπόν τη, τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την κατεξουσιοδότηση πράξη που εξετάζεται. Πριν πω στις λεπτομέρειες των ενστάσεων που έχουν εγερθεί και των θεμάτων που έχουν τεθεί σήμερα, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή και να σας θυμίσω το ιστορικό υπόβαθρο, πώς κατέληξε αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη να βρίσκεται ενώπιον σας σήμερα. Όπως είπε και η κυρία Γκέρλιν, πράγματι η πρόταση αυτή αποτελεί τη συνέχεια του 2013 και του κανονισμού που εκδόθηκε τότε για συγκεκριμένες διατροφικές ομάδες και τρόφιμα, όπου μέλη του Συμβουλίου, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασαν ιδιαίτερες ανησυχίες για την αύξηση των προβλημάτων ε, των υπέρβαρων και των παχύσαρκων ατόμων. Και δόθηκε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 να πράξει δύο πράγματα. Πρώτον, να ενημερώσει τους υφιστάμενους και ισχύοντες κανόνες που ισχύουν για τα προϊόντα ολικής υποκατάστασης γευμάτων Ε, με ε, περιεκτικότητα σε θερμίδες από 800 μέχρι 1200 ημερησίως και από, τη δεύτερη, από την άλλη πλευρά να ρυθμίσει ε, τα προϊόντα τα, με υπερβολικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες κάτω των 800 θερμίδων ημερησίως. Και για να το κάναμε αυτό και το κάναμε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, ήταν σημαντικό για εμάς να εκπληρώσουμε αυτό το στόχο. Δηλαδή να μεριμνήσουμε ότι όλα τα προϊόντα είναι κατάλληλα και ε, συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας. Και αυτό πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα και με την, ε, με σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις. Και γι' αυτό Διαβουλευτήκαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, είχαμε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας τροφίμων. Με το κοινό ερευνητικό κέντρο ε, κάναμε δουλειά πάνω στις τεχνικές ε, πτυχές για τα μεταποιημένα προϊόντα και τη διαδικασία ε, κατεργασίας και συσκευασίας αυτών. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι ε, ο κατεξουσιοδότης κανονισμός είναι η πιο κατάλληλη απάντηση στις ε, προσταγές σας του 2013 να ενημερώσουμε και να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες που διέπουν αυτά τα προϊόντα ολικής υποκατάστασης γευμάτων. Σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα με τα πρότυπα του κόντεξ του 95 σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για τη σύνθεση και τα συστατικά των, των προϊόντων σε ό,τι αφορά το κόστος και ε, τις απαγορεύσεις σε θέματα υγείας πιστεύουμε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Όλες αυτές τις διαστάσεις τις έχουμε εξετάσει. Ο κόντεξ του 1995 δεν αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις ε, της επιστήμης στον τομέα αυτό. Και ισχύει αποκλειστικά και μόνο σε προϊόντα με πολύ χαμηλή θερμιδική πρόσληψη που παρουσιάζονται με τη μορφή της φόρμουλας. Δεν είναι προϊόντα ολικής υποκατάστασης διατροφής, ούτε ούτε είναι τα προϊόντα των ε, ε, συστημάτων διατροφής πολύ χαμηλών ε, σε θερμίδες. Είναι μια υποκατηγορία αυτής της δεύτερης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση τα πρότυπα του 95 δεν έχουν διαμορφωθεί με βάση, τις πιο πρόσφατες, με βάση τα πιο πρόσφατα ευρήματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και εμεί θέλουμε να βασιζόμαστε σε αυτά. Σε ό,τι αφορά τα, τις προϋποθέσεις για τη σύνθεση των προϊόντων και τα συστατικά τους. Μας ενδιαφέρει κυρίως η ασφάλεια των καταναλωτών και ακολουθήσαμε την επιστημονική ε, σύμβουλη της ΕΦΣΑ έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά η ολικής υποκατάστασης να καταναλώνονται με ασφάλεια από υπέρβαρους και παχύσαρκους. Η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ασχολείται και υποκλειστικό της μέλημα είναι η ασφαλής κατανάλωση. Και γι' αυτό έχουμε την άποψή της ως σημείο εκκίνησης Και με το τεχνολογικό σκέλος θα ασχοληθούμε ξεκινώντας από τις ε, διαταγές της ΕΦΣΑ για το τι είναι ασφαλές να καταναλωθεί και τι όχι. Εξετάσαμε προσεκτικά τις επιστημονικές σύμβουλες και είδαμε κατά πόσο όλα αυτά είναι εφικτά από τεχνική σκοπιάς και κάναμε εκτεταμένη διαβούλευση με τους ε, ενδιαφερόμενους εταίρους. Δύο χρόνια κράτησαν αυτές οι διαβουλεύσεις από τότε που ε, κατέστη δημόσια η Επιστημονική Συμβουλή της ΕΦΣΑ. Η πρόταση ψηφίσματός σας εκφράσει ανησυχίες για τη μεθοδολογία που ακολούθησε η ΕΦΣΑ και για την τεχνική του ε, παίρνω κάποια δεδομένα που ισχύουν και τα αποδίδω την τεχνική των προβολών δηλαδή ε, των στοιχείων. Έχουμε την ημερήσια συνιστόμενη πρόσληψη για τους φυσιολογικούς εντός αγωγικών ενήλικες, κανονικού βάρους, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, θεωρεί η ΕΦΣΑ ότι είναι το ε, οι καλύτερες δυνατές προβλέψεις για να εκπροσωπηθεί και ο πληθυσμός των υπέρβαρων και των παχύσαρκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι ιδιαίτερη η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αλλά ακολουθήθηκε ακριβώς γι' αυτό, για να, έχουμε, να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των ανθρώπων και να ακολουθήσουμε στενότερα τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις. η ΕΦΣΑ αναγνωρίζει ότι η προσθήκη των απαραίτητων αυτών λιπαρών οξέων ενδεχομένως δεν χρειάζεται. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι υπάρχει ασάφεια ε, στο κατά πόσο τα, οι, οι αποθήκες σε του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος ε, για τους οργανισμούς, για τους ανθρώπους που ακολουθούν αυτού του είδους διατροφής επαρκούν για να είναι σε λιπαρά οξέα, δηλαδή για να είναι ισορροπημένη η διατροφή τους εξού και έχουμε προσθήκη των απαραίτητων λιπαρών οξέων. Σε κάθε περίπτωση τα επιστημονικά στοιχεία είναι πολύ καλά τεκμηρωμένα, αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Λάβαμε υπόψη μας τις τεχνικές πτυχές, Διαβουλευθήκαμε με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο για το θέμα αυτό. Είχαμε συναντήσεις με τους εταίρους και συνομιλητές μας και δεχθήκαμε και συμβουλές σε σχέση με τις τιμές που προτείνει η ΕΦΣΑ. Όλα αυτά τεχνολογικώς είναι εφικτά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ε, γίνεται και από τεχνικής και οικονομικής σκοπιάς να κατασκευάσει, να παρασκευάσει κανείς προϊόντα εύπεπτα που να μπορούν να κατανολωθούν με ασφάλεια. Το Σεπτέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο και τη Βιομηχανία όλες αυτές τις περίπλοκες τεχνικές πτυχές για τα προϊόντα ολικής υποκατάστασης Έχουμε την μικροκαψακίωση, δηλαδή το να περικλειστούν σε δισκία και σε κάψουλες τα στοιχεία. Υπάρχουν τεχνικές που καλύπτουν δηλαδή τις, ε, ε, τις ανησυχίες, τις καταλαγιάζουν, ειδικά τις ανησυχίες που έχουν να κάνουν με την οσμή αλλά και το εύγευστο ε, των προϊόντων. Πολλές συμβουλές δεχτήκαμε από πολλούς εταίρους. Σύμφωνα με τις δικές μας αξιολογήσεις, τα επιπρόσθετη κόστη δεν συνδέονται με το κόστος της πρωτεΐνης, αλλά με το κόστος της, του, της κατασκευής, του μάρκετινγκ, της διανομής. Και η αύξηση που εκτιμάται δεν είναι καθόλου σημαντική. Είναι πολύ μετριοπαθής η αύξηση του κόστους σύμφωνα με τις προβλέψεις μας. Δεν σας άκουσα κύριε Πρόεδρε, με διακόψετε. Α, θέλετε να ολοκληρώσω. Θα συντομεύσω. Τελευταία παρατήρηση. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο, το ενεργειακό είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συμβουλή ειδικού μέχρι 8 εβδομάδες μόνο είναι άποψη της ΕΦΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να τίθενται σε εμπορία με διαφημιστικά μηνύματα και ισχυρισμούς που ε, θα μπορούσαν να προσελκύσουν το σύνολο του πληθυσμού. Δεν το επιθυμούμε να υπάρχουν μηνύματα που προσελκύουν το σύνολο του πληθυσμού αφού θα απευθύνονται μόνο ε, στα ε, παχύσαρκα άτομα. Άλλωστε έχουμε και μια μεταβατική περίοδο των 5 ετών και πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την περίοδο θα ξεπεραστούν όλα τα τεχνολογικά εμπόδια, τα εμπόδια κατά τη μεταποίηση και θα είναι απρόσκοπτη η μετάβαση στη νέα κατάσταση όπου θα υπάρχει συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στο, στη συνεισηγήτρια για μια σύντομη αντίδραση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καταστήσω κάτι σαφές. Γιατί υπάρχει σύγχυση. Δεν ρυθμίζουμε κάτι καινούριο. Δεν είναι ένας νέος κανονισμός τον οποίο θέλω εγώ να καταργήσω. Υπάρχει κανονισμός. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ρυθμίζονται αυτά τα προϊόντα. Υπάρχει ήδη κανονισμός για αυτά τα προϊόντα. Έχουμε κάνει αλλαγές μεταξύ ενηλίκων και δεν διαφωνώ με τις περισσότερες αλλαγές. Και μάλιστα στις ενστάσεις μου καμία σχέση δεν έχει η σήμανση, η ετικετοθεσία και χαίρομαι ιδιαίτερω με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην υπάρχουν ισχυρισμοί υγείας δηλαδή για το σύνολο του πληθυσμού ε, σε όλη την ετικετοθεσία και τη σήμανση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι δεν έχει μια σχέση με αυτό. Η ένστασή μου έχει να κάνει με τη σύνθεση και με το εύπεπτο, το εύγευστο, το κατά πόσο μπορούν πραγματικά να τα φάει κανείς, να τα καταναλώσει αυτά τα προϊόντα. Νομίζω ότι λέμε στον κόσμο που χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα πολύ αποτελεσματικά και θέλω σε παρένθεση να πω ότι πολλούς τέτοιους συνάντησα πριν γύρω τις ενστάσεις μου δεν, έβαλα, δεν έγινε αυτή την έσταση γιατί στηρίζω τη βιομηχανία, αλλά γιατί είμαι υπέρ των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Και από όλες αυτές τις συναντήσεις, τις μακροσκελείς συνομιλίες που είχαμε τους καταναλωτές, κατάλαβα πόσο σημαντικά είναι αυτά τα προϊόντα για αυτούς, πόσο τεράστια διαφορά έκαναν και έφεραν αυτά τα προϊόντα στην υγεία των ανθρώπων αυτών και γι' αυτό ε, ε, έχω αυτές τις ενστάσεις για το εύγευστο και για τη δυνατότητα να ε, καταναλωθούν τελικά αν περάσουν οι νέες προϋποθέσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει λάθος ως προς το εύπιο το αν θέλετε το, ε, το να μπορούν να, ε, οι άνθρωποι να τα καταναλώσουν. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι θέμα δεξιάς και αριστεράς, δεν είναι θέμα του αν στηρίζει κανείς την Ευρωπαϊκή Μέθοδο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι. Είναι μια ένσταση πολύ συγκεκριμένη που έχει να κάνει με τη δυσκολία κατανάλωση αυτών των προϊόντων με τη νέα κατάσταση. Και αν υπάρξει καθυστέρηση, αυτό δεν είναι ενδεχομένω πρόβλημα. Πάντω μην νομίζετε ότι τα προϊόντα είναι αρρύθμιστα. Ήδη υπάγονται σε ρυθμίσει και προποθέσει με βάση τα πρότυπα του κόντεξ. Σα ευχαριστώ πολύ. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. περιμένετε να βγάλουμε τις κάρτες μας και τις λίστες ψηφοφορίας. Λοιπόν, μπορείτε να ψηφίσετε, ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό. Το επόμενο, προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Δύο ψηφοφορίες. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρα της ψηφοφορίες. Δεκτό. Η επόμενη ηλεκτρονική ψηφοφορία, πάλι προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτές. απαιτήσει για αντιρρήσει. Electronic vote. I open Για τα υποκατάστατα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 18 όλα τα τμήματα Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 3, αποχέ, δεκτό 4 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 10 υπέρ κατά αποχές απερίφη 9 υπέρ κατά αποχές απερίφη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφη 12 υπέρ κατά αποχές απερίφη 15 υπέρ κατά αποχές απερίφη 14 υπέρ κατά αποχές δεκτόι 13 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 16 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 18 υπέρ ή έχει καταπέσει μάλλον, ή 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ηλεκτρονική ψηφοφορία ή τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρα της ψηφοφορίας, δεκτή. Συγχαρητήρια λοιπόν Η επόμενη ψηφοφορία είναι η δημοσιονομική διαδικασία για το 18, τροπολογίες στον προπολογισμό. Θα διαβάζω τους αριθμούς. 147 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 5, 4, 44 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 5-4-4-8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5-4-4-9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5-4-10 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5-4-10. Τέλος. Δεκτή. 5-4-11 11 ειπε κατά αποχές απερίφθη 5-4-5-4 4 είπε. κατά αποχές δεκτή 5-4-12 μαζί με την 5-4-55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5-4-13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεκτή. 5456 και 5457 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 5458 και 5459 ομαδών υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 5460, 5461 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 62 και 63 συνολική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές δεκτές 54-36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54-64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-21 υπέρ κατά αποχές απερίφη 54-53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-22 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 54-46 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 54-14 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 54-15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 54-16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16. 26 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Ελέγχουμε την 54-26 ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφοριας απεριφη Απερίφθη. 54-27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54-29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-34 υπέρ κατά αποχές δεκτή απερίφη μάλλον, 54-35 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη, 54-28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 54-18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 54-45 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη, 54-88 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 54-24 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 54-23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5470 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5471 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5477 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5472 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5474 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54-38 υπέρ κατά αποχές απερίφη 54-40 υπέρ κατά αποχές απερίφη 54-41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54-43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 54-06 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 54-75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54.00 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 54.76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54.77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54.05 και 54.78 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές 5479 υπέρ κατά αποχές δεκτές 5404 υπέρ κατά αποχές απερίφη 5483 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5403 υπέρ κατά αποχές απερίφη 5402 υπέρ κατά αποχές απερίφη 5401 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5450 υπέρ κατά αποχές αδεκτή 5451 υπέρ κατά αποχές Ξανά παρακαλώ ποιοι είναι υπέρ της 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5452 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 54, 66, 67 και 68 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές δεκτές, 54, 80 και 81 υπέρ, α και 82 επίσης, τρεις τροπολογίες, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 54, 85, 86 και 87 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Αποχές ε, δεκτές. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54, 09 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54, 08 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Δίνω την Προεδρία τώρα πλέον στην κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ πολύ. S'il vous plaît, chers collègues, Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι για να συνεχίσουμε. Έχουμε καθυστερήσει κάπω. Οπότε, ευχαριστώ όσου παραμένουν στην αίθουσα. Περάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι το σημείο στην ημερήσια διάταξη για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας. Για να μην χάνουμε χρόνο, θα δώσω το λόγο αμέσως στην εισηγήτρια, που είναι η κυρία Μελά, από το ΙΕΝΕΦ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρόλο που έκθεσή μου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που έχουν να κάνουν σε έκθεση ε, καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων ουσιών απορρίφθηκε από τις περισσότερες ομάδες εδώ στην Επιτροπή μας. Παρόλα αυτά δεν είναι ένα θέμα πολιτικοποιημένο και έτσι όπως εξετάζω εγώ τη δεύτερη πτυχή δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία και την πολιτική. Διακόπτει ομιλήτρια. Στο ίδιο πνεύμα λοιπόν, ε, προστασία τη εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην αξιολόγηση των κινδύνων για του εργαζόμενου από τη μία και τη δυσκολία των επιχειρήσεων από την άλλη, να πώ θα φτάσουμε σε ένα μηδενικό κίνδυνο. Κύριε Πρόεδρε, λέει η ομιλήτρια, δεν θα συνεχίσω, θα περιμένω να έχουμε ησυχία για να μπορώ να μιλήσω. Πρόεδρος, Πράγματι δεν είμαστε τόσο πολλοί σε αυτή την αίθουσα. Παρακαλώ να κάνουμε όλη την προσπάθεια να μπορέσουμε να ακούσουμε την εισηγήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, έλεγα ότι στο ίδιο πνεύμα τη προστασία τη ισορροπία αυτή ανάμεσα στου κινδύνους για την υγεία από τη μία και την προσπάθεια των επιχειρήσεων να φτάσουν μηδενικό κίνδυνο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, καταλήγω στην πρότασή μου για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερο και που έχει να κάνει με όλες τις χώρες. Θα εξετάσω με ανοιχτό πνεύμα όλες τις τροπολογίες που θα φτάσουν, λέγοντας ότι προσωπικά, πέρα από τα παραρτήματα, δεν τροποποίησα το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τολμάω να πιστέψω ότι συνάδελφοι από την Επιτροπή αυτή περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας θα μπορέσουν για δεύτερη φορά να οδηγήσουν σε αφαίρεση κάθε νομιμότητας. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι δέχονται τις ρυθμίσεις εφόσον αυτές έχουν προηγουμένως συζητηθεί επαρκώς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι σκιώδες που απουσιάζουν σήμερα, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέριγκερ από το ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των εργαζομένων φυσικά και πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας. Δεν είναι δυνατόν να θυσιάζουμε την υγεία των ανθρώπων πρέπει να ξέρουμε ότι οι υγιείς άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί, άρα ευνοούν και την παραγωγικότητα. Οπότε η πρόταση επιτροπής είναι μια πρόταση από την οποία όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όλοι. Η καλή πολιτική είναι και η δύναμή μας στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη κοινομοδότηση. ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο της. Οι νέες οριακές τιμές πρέπει να είναι εφικτές και μετρήσιμες. Όμως η ομάδα μου στηρίζει τις οριακές τιμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε μια επιστημονική διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή για να καταλήξει σε αυτές τις οριακές τιμές. Συνεπώς έχουμε τάση να μην συμφωνήσουμε στις αλλαγές που προτείνει η συγγήτρια στη γνωμοδότηση. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες οι οποίες θα καταδεικνύουν και τη θέση μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Στην αίθουσα έχουμε ακόμα τον κύριο Έικ. Είναι σκιώδης για την ομάδα του. Παρακαλώ κύριε Έικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ασφαλώς και πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι επιτέλους έχουμε μια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας που αναφέρεται στην έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες είναι κάτι που έχει ανακοινωθεί εδώ και χρόνια. Η Επιτροπή καθυστέρησε επειδή έπρεπε να τηρηθούν διάφοροι κανόνες για την καλύτερη νομοθέτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θέλει να προστατεύσει τους εργαζόμενους από τις επικίνδυνες αυτές ουσίες και η βιομηχανία από την πλευρά της είναι αλήθεια ότι δεν θα πρέπει να υποβληθεί σε περιορισμούς, συμφωνούμε. Όμως ο καρκίνος παραμένει να είναι η πρώτη αιτία θανάτων στην Ευρώπη σήμερα. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πρόληψης πρώτα απ' όλα από τη βιομηχανία. Νομίζω λοιπόν ότι η αρχή αυτή πρέπει να τηρηθεί και συχνά την έχουμε ξεχάσει. Όλα αυτά είναι του παρελθόντος. Χαιρετίζω λοιπόν τις πιο αυστηρές διατάξεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, αλλά λυπούμε που κάποιες ουσίες δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις επί της γονιμότητας. Θα έπρεπε λοιπόν επίση οι ενδοκρινικοί διαταράχτε να συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση αυτή. Ζητάω από την Επιτροπή να το λάβει υπόψη τη. και να καλύψουμε επίση και άλλα τοξικά στοιχεία. Να μην περιοριζόμαστε σε ουσίε γιατί δεν πρόκειται μόνο για του εργαζόμενου, αλλά πρόκειται και για τα παιδιά που θα γεννήσουν αυτοί. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Τώρα, ο συνάδελφος Πεντιτσίνη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μένοντας δεδομένα στα στοιχεία που βλέπω στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα οποία δεν μπορώ να αμφιβάλλω, βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλός αριθμός ε, συχνές περιπτώσεις ε, δημιουργίας προβλημάτων υγείας καρτίνου λόγω ακριβώς ε, της έκθεσης σε παραγωγή προϊόντων καρκινογόνων και ανάμεσα σε αυτά το 57% των 100.000 δυστυχώς οδηγούν στο θάνατο των ασθενών. Συνεπώς λοιπόν βλέπουμε ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε σε καθημερινή βάση 37 τουλάχιστον θανάτους από τον καρκίνο που οφείλεται σε επαγγελματικές αιτίε. Πρέπει να το καταπολεμήσουμε λοιπόν με αποφασιστικότητα. Συμφωνούμε πλήρως λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη βάση της αξιολόγησης των επιπτώσεων. Θέλει να μειώσει την έκθεση των εργαζομένων. Δεν περίμενα από την Επιτροπή μας να προτείνει κάτι το οποίο θα ήταν ασθενέστερο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να υπενθυμίσω στην εισηγήτρια ότι η έκθεση στις καρκινογόνες ουσίες δημιουργεί, αν θέλετε, έκθεση, δυνατότητα έκθεση σε κίνδυνο, ακόμα και με ε, πολύ λίγες πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν τα όρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούνται ιδιαίτερα αυστηρά από την εισηγήτρια ε, για την βιομηχανία, τότε θα πρέπει η βιομηχανία η ίδια να βρει εναλλακτικέ ε, λύσεις με μηδενικό κίνδυνο για τους εργαζομένους. Εμείς λέμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος των εναλλακτικών και όχι ο εργαζόμενος ο οποίος κινδυνεύει να ασθενήσει. Ακόμα και αν υπάρχει κίνδυνος έστω και για ένα μόνο εργαζόμενο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελαν το λόγο για την έκθεση Μελάν. Δεν υπάρχει κάτι. Θα στραφώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εισηγήτρια κυρία Ζωέρ Μελάν για την γρήγορη αντίδρασή σα την οποία εκτιμούμε δεόντως, διότι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και εμείς τη δουλειά μας γρηγορότερα. Η προστασία των εργαζομένων είναι εξόχω σημαντική. Αυτή η δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με αυτά που προτείναμε το Μάιο θα βοηθήσει να σώσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές τα επόμενα 50 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ως προς το σχέδιο γνωμοδότησης, και τις προτάσεις να αυξηθούν οι τιμές στον εργοσιακό χώρο, να σας πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία τα οποία στα οποία έχει καταλήξει η επιστημονική μας επιτροπή. Έχουμε κάνει αξιολόγηση επιπτώσεων αντικτύπου, έχουμε εξετάσει τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές, το κατά πόσο όλα αυτά είναι τεχνολογικώς εφικτά και για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κάναμε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και είχαμε και τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι τιμές είναι εφικτές και μπορεί να εφαρμοστούν. Ως προς το σχόλιο του κυρίου Εκ, Εκ για τις ουσίες αυτές, με την πρώτη τροπολογία της οδηγίας CMD είχαμε φτάσει σε συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει το ζήτημα και η αξιολόγηση θα είναι έτοιμη το 2019. Θα σας ευχαριστώ όλους για την αδεία συνεργασία και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ για τα συμπεράσματα να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μίλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λαμβανώντας υπόψη το πόσο γρήγορες ήταν αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες ήταν κάπως αναξιοπρεπής θα έλεγα, ε, με δεδομένη τη σοβαρότητα και την περιπλοκότητα της κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν να, να υπογραμμίσουμε εδώ κάποιες πτυχές πολύ σημαντικές που μπορεί να μην υπάρχουν στους φακέλους. Όταν όμως ολοκληρώνουμε τις υποθέσεις, θα πρέπει οι εργαζόμενοι που πάσχουν από κάποια νόσο να μπορούν να την αποδώσουν όταν αυτόν ισχύει ε, με την εργασία την οποία έκανα προηγουμένως. Διάφορα ε, νοσήματα έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Οφείλονται, είναι πολυποραγοντικά δηλαδή. Και είναι πολύ δύσκολο κανείς κατηγορηματικά να πει ότι ο αμύαντος και όχι το κάδμιο και όχι κάποιο άλλο χύψη προϊόν έχει άμεση σχέση με την εκάστοτε νόσο, με το εκάστοτε νόσημα που εμφάνισε ο ασθενής. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, οι εργαζόμενοι μετακινούνται, μετεγκαθίστανται. Πώς θα το κάνουμε. Έχουμε, ακόμα και αν έχουμε ταυτόσιμες τιμές ανώτατης έκθεσης των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παράγοντα, ε, όταν άνθρωποι 60, π.χ. 65 ετών παρουσιάζουν καρκίνο πνεύμονα που έχει άμεση σχέση με την έκθεση σε χή παράγοντα, σε χή χώρα, σε χή επιχείρηση, πώς θα το αποδώσουμε σε αυτό όταν το άτομο έχει ασκήσει τα καθήκοντά του σε διαφορετική χώρα και σε διαφορετικό τομέα. Κύριε Πεντιτσίνη, στην επαγγελματική μου ζωή έχω ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που είναι θύματα εργασιακών ασθενειών. Πώς ε, θα φροντίσουμε καλύτερα τα συμφέροντά τους. Κάποιες τιμές έκθεσης ανώτατες δεν μπορούν να ισχύσουν σε κάποιες χώρες, είναι ανεφάρμοστες. Πώς θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ των μεν ούτε υπέρ των δε. 40 χρόνια έχω εργαστεί με απόλυτη ουδετερότητα και σήμερα είμαι εδώ παρούσα με απόλυτη οικονομική, πολιτική αλλά και φιλοσοφική ουδετερότητα. Βρίσκομαι εδώ για τη διατήρηση των θέσεων απασχόληση σε καλέ συνθήκε εργασία να είναι αυτό εφικτό για του εργαζομένου και να προστατεύονται και εργαζόμενοι και εργοδότε. και χαίρομαι διότι υπάρχει η αρχή τη προφύλαξη και υπάρχει αυτό στην πρώτη υπόθεση, στο πρώτο φάκελο, η αρχή τη προφύλαξη και επιθυμώ με αυτό να διατηρηθεί και γι' αυτό υπέβαλα δέκα τραπολογίε σε αυτή την πρώτη έκθεση που δεν έγιναν δεκτές, ε, απορρίφθηκαν όλες. Τα κράτη και οι εργοδότε είναι αυτοί που πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε υποκατάστατα και να εξαφανιστεί ο καρκινογόνος παράγοντας. Είναι πολύ εύθραυστη αυτή η ισορροπία να είμαστε και αποτελεσματικοί και να είναι εφαρμοστέα, να μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που προβλέπουμε. Με μεγάλη χαρά θα παραστώ σε συνάντηση με σκιώδους εισηγητές. Με για να ανταλλάξουμε υπόψεις για τις τροπολογίες. Ε, θα ήθελα όλοι να μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ε, δεχθώ τις τροπολογίες ελπίζοντας να γίνει δεκτή και η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, να σας υπενθυμίσω κάποιες βασικές ημερομηνίες. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. 6 Σεπτεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας για το περιβάλλον στις 12 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή για την Απασχόληση 27 Νοεμβρίου και δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 11 στην εμμυρίσια διάταξη. Πρόκειται για το, πρόγραμμα, το σχέδιο δράσης για τη φύση, των άνθρωπο και την οικονομία. Και θα δώσω το λόγο στους διάφορους συνεισηγητές. Πρώτα απ' όλα στον συνάδελφο Ντόρφαν, εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ψηφίσαμε την προφορική ερώτηση πριν και η συζήτηση έχει τώρα να κάνει με το ψήφισμα. Καταρχήν, εκ μέρους της ομάδας μου, μπορώ να πω ότι φυσικά και στηρίζουμε το Natura 2000, τη βιοπικιλότητα, είναι πράγματα με τα οποία ασχολείται πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βιοπικιλότητα στην Ευρώπη δεν έχει να κάνει μόνο με τα τοπία, έχει να κάνει και με τη γεωργία. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τη δράση του ανθρώπου και να πετύχουμε μια ισορροπία έτσι ώστε να σεβόμαστε τη φύση. Ακριβώς λοιπόν οι περιοχές Natura 2000 έχουν οδηγήσει σε κάποιες συγκρούσεις οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Πρόκειται για ευαίσθητες περιοχές όπου η ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό τοπίο και την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολύ ευαίσθητη. Κυρίως ε, μάλιστα στις περιοχές από όπου προέρχομαι εγώ. Αυτό που θέλω εδώ να καταδείξω είναι ότι το ζήτημα σαρκοφάγων όπως είναι ο λύκος, ε, η αρκούδα έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πολεμική. Και στο ψήφισμα αναγκάστηκα να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα από τη μια στην αναγκαιότητα να προστατεύσουμε την παραδοσιακή γεωργία και από την άλλη το γεγονός ότι οι λύκοι για παράδειγμα μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε κάτι το οποίο θα έχει αρνητικές συνέπειες, γιατί η παραδοσιακή γεωργία ε, θα χαθεί. Τα λιβάδια, ας πούμε, στις Άλπεις. Πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό το ζήτημα, πόσο δηλαδή θα καταλήξουμε σε μια λογική λύση, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη ανάμεσα στα μεγάλα σαρκοφόγα και τις ανάγκες της γεωργίας κυρίως της Άλπης. Να δούμε ποια είναι τα επιπλέον μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία. Αυτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, κύριε Κάτεπαχ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ντόρφμαν είπε κάποια πράγματα που θέλουμε και εμείς να δούμε στο ψήφισμα αυτό. Ε, για παράδειγμα, πρέπει να αναφέρουμε ότι για να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα ε, πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι τομείς, όλες οι πλευρές. Ο άνθρωπος, η φύση, η οικονομία. Οι μισές επιφάνειες Natura 2000 δεν είναι στη διάθεση του ανθρώπου για να κάνει χωροταξιακό προγραμματισμό και υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία μπορούν να επιβιώσουν βέβαια σε αυτές τις περιοχές χωρίς όμως να έχουμε πετύχει απόλυτα το στόχο μας ακόμα. Χρειάζεται καλύτερη ισορροπία Αναφέρθηκε η σύγκρουση από τον κύριο Ντόρφμαν που διαπιστώνεται μερικές φορές. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε και το θέμα των προστατευόμενων ειδών. Τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές υπάρχει κίνδυνος για σύγκρουση εάν η ιδιοπικιλότητα παρουσιάζεται πιο περίπλοκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν πληθυσμοί που εκπροσωπούνται υπερβολικά και πρέπει να τους προστατεύσουμε. Η λύση στην οποία θα καταλήξουμε πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη. Που να λαμβάνει υπόψη και τη γεωργία και τη δασοκομεία. Χρειάζεται ελαστικότητα, χωρίς βέβαια να τίθεται σε κίνδυνο οι κανόνες προστασίας. Αναφέρθηκαν η Αρκούδα και ο Λύκος και νομίζω ότι ότως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε επαόριστο. Η προστασία των ειδών, η βιοπικιλότητα είναι πράγματα τα οποία θα πετύχουν εφόσον ο πληθυσμός είναι πεπισμένος για την αναγκαιότητα αυτής της συνύπαρξης των διαφορετικών ειδών. Πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη. Θα το πετύχουμε μακροπρόθεσμα αν μας στηρίξει ο κόσμος. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με την Αρκούδα και το Λύκο. Βλέπουμε ότι οι Λύκοι έχουν μετακινηθεί και κυκλοφορούν ευρύτερα. Μερικές φορές μάλιστα υπάρχουν και υβριδικές μορφές λύκων επειδή συνεπάρχουν με τα σκυλιά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί να λάβουμε υπόψη μας αυτή την κατάσταση. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για να καταλήξουμε σε μια λύση που να καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα. Πιο αποφασιστικά ακόμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρους του ECR, ο κύριος Τεσμάκερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, συζητήσαμε την έκθεση για την βιοπικιλότητα που εγκρίθηκε και ένα από τα βασικά μηνύματα στην έκθεση αυτή ήταν ότι η απώλεια βιοπικιλότητας πρέπει να σταματήσει και ότι πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα αυτό. Η προστασία δηλαδή της βιοπικιλότητας είναι κάτι αναγκαίο, απαραίτητο και για την φύση, αλλά όχι μόνο για τη φύση, αλλά και για τη δικιά μας την ευημερία και τη δικιά μας την ε, ύπαρξη και την οικονομία ακόμα. Έχουμε τους, τους στόχους του 2020. Αναφέρεται και η προστασία της φύσης και είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές που δεν θα τροποποιήσει στη συνέχεια. Το πρόγραμμα δράσης τώρα πρέπει βέβαια να φροντίσει πιο γρήγορα να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Συγχρόνως όμως πρέπει να πετύχουμε τους στόχους του 2020, άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια. Και αυτό φάνηκε και τον Ιούνιο από την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μας λοιπόν περιβάλλοντος πρέπει να στείλει ένα μήνυμα για το τι μπορεί να γίνει καλύτερα και τι πρέπει να γίνει καλύτερα. Και το ψήφισμα που έχουμε μπροστά μας ακριβώς αναφέρει τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχέδιο δράσης. το σχέδιο δράσης δείχνει ότι δεν φτάνουν όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτευθούν οι στόχοι του 2020. Φυσικά με τη συμμετοχή όλων των διαφερομένων. Το σχέδιο δράσης επίσης αναφέρεται για την περίοδο μέχρι το 2020. Το μετά το 2020 όμως είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει στρατηγικό ε, σχέδιο και χρηματοδότηση. Και τέλος, το σχέδιο δράσης δεν απαντάει σε προκλήσεις όπως είναι η δημιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου πράσινων υποδομών. Πρέπει να γίνει αυτό για να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα τα διάφορα συμφέροντα, τη γεωργία, τη φύση, τη φύση, τη συνοχή κλπ. Είμαι ικανοποιημένο με το κείμενο που έχουμε μπροστά μας και ελπίζω να υπάρξει ευρεία στήριξη από αυτού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος Γκερμπραντή, εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα μπορούσα να επαναλάβω λέξη προς λέξη τόσα είπε ο συνάδελφος της Μάρκετ μόλις τώρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα, 100% μαζί του. Ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση είναι γιατί χάνουμε χρόνο. Ήμασταν στο κόκκινο σε όλα, μετά την έκθεση πριν από δύο χρόνια για τη φύση, και το σχέδιο δράσης τώρα είναι ένα καλό βήμα προς τα μπρος. Δεν θα φτάσει όμως για να αλλάξουν για αυτά τα κόκκινα φανάρια που είχαμε, που ήμασταν στο κόκκινο, τώρα να βρεθούμε στο πράσινο. και ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε να δραστηριοποιείται περισσότερο. Θεωρούμε ότι όλα τα άλλα συμφέροντα είναι πιο σημαντικά από εκείνο της φύσης, που έχει τεράστια όμως σημασία και για την ίδια αλλά και για μας το ανθρώπινο είδος. Ελπίζω λοιπόν ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επικεντρωθούμε σε αυτό το βασικό ζήτημα. Συμφωνώ ότι έχουμε πρόβλημα με κάποια είδη, και έχει νόημα να τα αναφέρουμε και αυτά. Το κύριο πρόβλημα όμως δεν είναι η λύκη που εμφανίζονται σε κάποια σημεία της Ευρώπης ή κάποια άλλα είδη αλλού. Το θέμα είναι χιλιάδες χιλιάδων είδη τα οποία απειλούνται σήμερα. Και αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό μας σημείο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ότι και η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα θα καταλήξει σε αλλαγή νοοτροπία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για ένα σχέδιο δράσης μέχρι το 2020. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ιδίως σε εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην γεωργική πολιτική, ο Επίτροπος Χόγκαν δεν μπορεί να ξεφύγει λέγοντας ας περιμένουμε την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Όχι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ανοιχτά να πει συγγνώμη, δεν θα τα έχουμε καταφέρει με τη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα για το 2020. Για μένα λοιπόν, πολιτικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Να επικεντρωθούμε στα βασικά ζητήματα που δεν καταφέρνουμε να καλύψουμε με την πολιτική μας για την βιοπικιλότητα στην Ευρώπη και να κάνουμε κάτι παραπάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Οι υπόλοιποι συνεισηγητές δεν είναι παρόντες εδώ, οπότε έτσι θα περάσουμε στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Χέλνερ είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Ένα θέμα θα ήθελα να θέσω για την βιοπικιλότητα και την πολιτική μας γύρω από αυτή. Να αναφερθώ στις οδηγίες για τα πτηνά και το περιβάλλον. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Γκιομπράντη, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον πέρα από το πήγαινε έλα στο Στρασβούργο το οποίο δεν καταλαβαίνουν οι εκλογέ μου είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της βιοπικιλότητας στην οδηγία Habitat και στην οδηγία για τα πουλιά. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να με βοηθήσετε έτσι ώστε να μπορέσω να δώσω ε, μια ικανοποιητική εξήγηση για αυτό το οποίο συμβαίνει. Διαρωτώ με λοιπόν αν θα μπορούσε να το κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ε, πάει κανείς στην Στοκόλμη και σε άλλα μέρη της Βαλτικής ε, και βλέπει ε, κυρίως... Speak to people and they say they've been exploding, uh, but you're not allowed to hunt them because Εν πάση περιπτώσει το μόνο που βλέπει είναι ένα είδος ε, ε, από πουλιά και όχι πια ε, πολλούς γλάρους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα αλλιεύματα έτσι και αλλιώς στην Βαλτική. Αυτό μπορεί να συνδέεται και με την επιβίωση των, της ποικιλία, της βιοπικιλότητας στην, στα πουλιά. Ε, θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά εκδίδοντας μόνο άδειε αποκλήσεων. Άδειε αποκλήσεων είναι εξαιρέσεις ουσιαστικά από την νομοθεσία. Και η εμπειρία των Σουηδών πολιτών δείχνει ε, ότι δεν είχαμε πάντα επιτυχία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ε, είχαμε οδηγήσει τους λύκους, σαν παράδειγμα, να κυκλοφορούν στα περίχωρα της Ουψάλα ελεύθεροι σε κάποια φάση. Συνεπώς λοιπόν έπρεπε να ζητήσουμε μια εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τους λύκους η λογική που λέει ότι δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα είδη και γενικότερα στη βιοπικιλότητα γενικότερα είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά και δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί τους, ε, ε τους πολίτες. Γιατί τα διάφορα είδη στην, ε, στο παρελθόν υφίσταντο διαφορετικού τύπου πιέσεις από ό,τι σήμερα. Η κατάσταση με τους λύκους σήμερα στη Σουηδία είναι εντελώς διαφορετική από ότι ε, στο παρελθόν, από ότι 15 ε, χρόνια. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιοποικιλότητας γενικότερα. Νομίζω ότι οι οδηγίες αυτές έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί δεν είναι αποτελεσματικές. Έχουμε κάποιους στατικούς καταλόγους των ζώων σε όλες τις οδηγίες που δεν αλλάζουμε, ενώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυναμική στο περιβάλλον, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει συνεχώς. Συνεπώς, λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλησε να προχωρήσει ε, σε αναθεωρήσεις των καταλόγων. Φοβάμαι ότι με τα στοιχεία τα οποία έχουμε πλέον στη διάθεσή μας οι ρυθμίσεις μας είναι αναποτελεσματικές. Προφανώς δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Στρασβούργο και από που πήγαινε ερχόμαστε στο Στρασβούργο, αλλά προσπαθήστε να μας εξηγήσετε ε, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα σε σχέση με συγκεκριμένες ποικιλίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια κάποια πρόταση. Θα ξεκινήσω με το Μαντέλα, αν και ακούγεται λίγο περίεργο. Εγώ ε, ε, είχα απασχοληθεί με το κίνημα εναντίον του Απαρτχάιντ και η φυσιογνωμία του Μαντέλα έδειχνε στο κοινό ότι υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι ε, στην Αφρική αλλά ο Μαντέλα ήταν ο πιο γνωστός και προκαλούσε την προσοχή και χρησιμοποίησαμε το μεμονωμένο πρόσωπο του Μαντέλα με το οποίο μπορούσε να ταυτιστεί ο πολίτης ενώ ε, δεν ήταν ο, ο μοναδικός πολιτικός κρατούμενος και ενδιαφέρθηκε το κοινό ε, και για τους υπόλοιπους. Ε, σαν παράδειγμα γίνεται μια συζήτηση για τους λίγκες και τις αγριόγατες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν γίνει προτάσεις έτσι ώστε στα σύνορα με τη Σκοτία να υπάρξει επανεισαγωγή από την ε, υπηρετική Ευρώπη της αγριόγατας ή λίγα για να υπάρξει αποκατάσταση του πληθυσμού. Ξέρω πως αντιμετωπίζονται ε, τα θέματα αυτά από το κοινό, Οι λύκη σαν παράδειγμα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που συγκεντρώνουν την προσοχή του κοινού Υπάρχει επίσης ε, και το θέμα των, ε, της αγριόγατας η οποία και αυτή σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης προκαλεί την προσοχή και ευαισθητοποιεί ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να κρατήσουμε όμως την ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς που ζητούν την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών βλαβών και ε, τους γεωργούς σαν παράδειγμα και θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές και δυστυχώς ε, οι αγρότες ε, στην βορειοανατολική Αγγλία ανησυχούν για τον πληθυσμό των προβάτων τους και των εγωιδών τους, αν υπάρξει επανεισαγωγή της άγριας γάτας. Ξέρουμε επίσης τι γίνεται και με τα ελάφια, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους πλέον και πολλές φορές πληρώνουμε ε, συγκεκριμένους κυνηγούς για να μειώσουν σε περιοχές με μεγάλη επιβάρυνση τους αριθμούς των ελαφιών. Ενώ κάποια ζώα ε, τα οποία αν υπανισαχθούν όπως ο λύκος ή η αγριόγατα μπορούν να το κάνουν αυτό από μόνα τους με φυσιολογικό τρόπο και μπορεί να βοηθήσει ε, ίσως ε, την αποκατάσταση γενικότερα της φυσικής ισορροπίας ε, ξέρετε ότι ακόμα και όταν φυτεύονται νέα δάση, τα δάση αυτά δυστυχώς πάρα πολύ νωρίς το πρωί στα μικρά δέντρα έρχονται τα ελάφια τα οποία ζουν σε πολύ μεγάλους πλέον πληθυσμούς και τα καταστρέφουν ε, τρώγοντας τα φύλλα της κορυφής. Και γι' αυτό λοιπόν ίσως η συζήτηση για τις αγριόγατες να είναι μια συζήτηση η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει ε, τη συνειδητοποίηση των προβλημάτων στα οποία μας οδηγεί η απώλεια της βιοπικιλότητας τις τελευταίες δεκαετίες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπέρντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε ότι το περιβάλλον αλλάζει. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περιβάλλον, έχει περιβάλλον το οποίο όχι μόνο αλλάζει αλλά επιδεινώνεται. Η αλλαγή είναι προς το χειρότερο, δεν είναι προς το καλύτερο ποτέ. Έχουμε τρία-τέσσερα project μόνο, το πολύ πέντε, που να βελτιώνουν τη βιοπικιλότητα σε όλη την Ευρώπη. Απειροελάχιστα δηλαδή. Όλη η φύση βρίσκεται υπό τεράστιες απειλές. Η βιοπικιλότητα συνδέεται με τις απειλές, με το ότι ε, ό,τι συμβαίνει σε ένα μέρος θα έχει σιωπηρές αρνητικές επιπτώσεις σε κάποια άλλη τοποθεσία. Αυτή είναι η λανθάνουσα σιωπηλή κρίση. Νομίζω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να προβλέψουν ένα διήμερο, να πάνε στον τόπο που μέναν όταν πηγαίναν στο δημοτικό. Αν επιστρέψουν στη γενέτειρά τους λοιπόν και δουν τι έχει εξαφανιστεί εκεί από την τότε τους γειτονιά, όταν περπατούσαν για να πάνε στο σχόλιο, τότε θα καταλάβουν τι έχει εξαφανιστεί στην προσωπική του ζωή. Γιατί εκεί έμαθαν τον κόσμο και εκεί ήταν η φύση πως είναι για πρώτη φορά. Αν πάνε σήμερα, όπου και αν είναι αυτό, σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο. Μόνο έτσι συνειδητοποιεί κανείς τις τεράστιες απώλειες. Και ε, πέρσι είχαμε μια εξαιρετική έκθεση για το θέμα αυτό και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για το μέρος της βιοποικιλότητας που χάνεται ανεπανόρθωτα. Και σε σχέση με τις συνδέσεις με άλλους τομείς πολιτικής και με αυτή την επικεφαλίδα, ένα από τα πολλά όνειδη θα έλεγα, ένα, ένα όνειδος της κοινή γεωργικής πολιτικής και μία από τις πολλές της αποτυχίες είναι η εξή ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν προστατεύει τα βοσκοτόπια. Υπάρχουν τοποθεσίες πολύ σημαντικές και πολύ ευάλωτες που είναι βοσκοτόπια και είναι πολύ ευάλωτα στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην, στην ε, Βουλγαρία, στην Πορτογαλία αλλά και στην Νοτιοανατολική Αγγλία αν θέλετε. Όλα αυτά ε, δεν προστατεύονται από την κοινή γεωργική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικά, όπως και οι αλπικές περιοχές. Έχουμε πανάρχια δέντρα σε αυτές τις τοποθεσίες που προστατεύονται από τον τρόπο ζωής και τον τρόπο καλλιέργειας και κτηνοτροφίας. Είναι σκληρή ζωή για τους κτηνοτρόφους, αλλά επειδή είναι ήπια η δραστηριότητα προστατεύεται πλειάδα ε, φυτικών και ζωικών ειδών. Πολύ σπάνια τα σχέδια τελικά εφαρμόζονται με τον επιθυμητό τρόπο. Και αν δεν έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για τα φωσκοτόπια τότε δεν θα τύχουν καμία απολύτω προστασία. Και αυτό θα έχει επιπτώσει και σε άλλου κρίκου τη αλυσίδα. Ο πληθυσμό που διαβεί εκεί μπορεί να ζει σκληρή ζωή, αλλά έχει πάρα πολλά ωφέλη, πολλέ χαρέ από τον παραδοσιακό τρόπο και την επαφή με τη φύση. Ε, ε, με τον πειμενικό αυτό τρόπο ε, ζωής. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό τον τρόπο ζωής και ε, να προστατεύσουμε τα ζωικά και φυτικά είδη που τους περιβάλλω. Όλα αυτά είναι εφικτά με σχεδιασμό, με χρηματοδότηση, με μέτρα όπως το σχέδιο δράσης που έχουμε. Εξού και υποβάλλω αυτή την τροπολογία. Ε, και κάποιες άλλες. Ελπίζω λοιπόν να μην ε, παραμελήσουμε τα βοσκοτόπια της περιοχής κτηνοτροφίας, φυσικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας και των ωφελιών για, όλου για όλους μας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, μετά από την παρέμβασή σας είναι η πολύ σημαντική άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Νοτάρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθυνθεί στην Επιτροπή σας και να αντιδράσει σε αυτό το ε, σχέδιο ψηφίσματος και τη συζήτηση που μόλις έγινε. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια στοιχεία και να πω ότι το σχέδιο δράσης και παραθετικά να πω ότι ευχαριστώ βεβαίω την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις θετικές της αντιδράσεις και ε, τη συμπερίληψη των ιδεών μας στο σχέδιο ψηφίσματος. Σε κάθε περίπτωση κλείνω την παρένθεση και λέω ότι το σχέδιο δράσης δεν είναι υποκατάστατο της ε, στρατηγικής για την βιοποικιλότητα, δεν την αντικαθιστά. Θέλει να διευκολύνει ε, την επίτευξη αυτών των στόχων. Βεβαίως υπάρχουν περιορισμοί και τους αναγνωρίζει το σχέδιο δράσης. Άλλωστε το χρονικό εύρος εκτείνεται μέχρι τη λήξη της θητείας της υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή μέχρι το 2019 θελήσαμε να υπάρχει λόγοδοσία για το, ε, ε, για το κατά πόσο θα επιτευχθούν οι δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης. Και θέλουμε μέχρι το 2019 να είμαστε σε θέση να δείξουμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε. Το σχέδιο δράση δεν μπορεί να προδικάσει ευρύτερε συζητήσει όπω είναι η συζήτηση για το μέλλον τη κοινή γεωργικής Πολιτική, η συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί την πρώτη συζήτηση του Κοινοβουλίου έχει τρομακτικό ρόλο, αφού είναι συνομοθέτη και συναποφασίζουν για το προπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση ε, όλα αυτά τα έχουμε τονίσει στην επικοινωνιακή διαχείριση του σχεδίου δράση. Μπορεί να συμβάλλει σημαντικά το σχέδιο δράση, Να πλησιάσουμε τους στόχους ε, της στρατηγικής βιοπικιλότητας για το 2020. Ε, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι ε, η οδηγία για τους βιοτόπους και για τα πτηνά δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό. Η βιοπικιλότητα έχει τεράστιο δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Έχουμε 1500 υποδράσει μεταξύ των βασικών δράσεων και ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται αρμονικά για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κανείς σήμερα δεν μπορεί να πει το κατά πόσο θα τα καταφέρουμε και αν ναι σε τι βαθμό, αλλά σε κάθε περίπτωση όλες οι προσπάθειες, όλοι οι πόροι έχουν σύστρατευθεί για να πλησιάσουμε το προσδοκόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή Επίσης, ορισμένες πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο σχέδιο ε, ψηφίσματος, όπως οι επικονιαστές για παράδειγμα και άλλα θέματα. Ξέρουμε τη σταυροφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία όλων αυτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές ε, ε, δεν έχουν επικυρωθεί πολιτικά. Εκρεμεί αυτό εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πολιτικό πράσινο φως, αλλά έχει γίνει προπαρασκευαστική δουλειά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλούμε επίσης για την λαθροθυρία ε, πτηνών και έχουμε ε, οδικό χάρτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λύσουμε το πρόβλημα. Συνομιλούμε με διάφορες οργανώσεις και εθνικές αρχές και την Ιντερπόλ και σε διεθνές επίπεδο και σε χώριο επίπεδο βασιζόμαστε στις διάφορες διεθνείς συμβάσεις για τα αποδημητικά μεταναστευτικά είδη, ε, ε, ε, συμβάσεις για την προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, διεθνείς συνθήκες που εκτείνονται και στην Ευρώπη και στην, Αφρο... και στην Αφρική. Σε κάθε περίπτωση δεν Είμαστε υπέρ της εισαγωγής των ειδών εκεί που έχουν εξαφανιστεί. Είναι ιδιαίτερη η περίπτωση του λύκου και η φυσική του αποκατάσταση σε βιοτόπους όπου είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν. Το καθεστώς προστασίας είναι που διευκόλυνε την ανάκαμψη των αποθεμάτων του ζωικού κεφαλαίου των λύκων. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Η αρχή στην οποία αναφερθήκατε κατοχυρώνεται στην οδηγία δεν γίνεται πλήρως αντιληπτή και κατανοητή και αξιοποιήσιμη και γι' αυτό το σχέδιο δράσης έχει προβλέψει συγκεκριμένες δράσεις για να υπάρχει περισσότερη ευελιξία, για χρήσεις περισσότερο κατανοητές, για να λυθούν οι συγκρούσεις μεταξύ ε, της προστασίας ειδών ε, που τα είδη έρχονται ε, σε σύγκρουση μεταξύ τους. Η προστασία και η άνθηση ενός είδους υπονομεύει την επιβίωση κάποιου άλλου. Μιλούμε για περίπου 10 είδη που ίσως ε, δημιουργούν κάποιες εντάσεις από τα 1500 είδη που προστατεύονται στην Ευρώπη. Μόνο για ε, περίπου 10 γίνεται ο λόγος. Ε, πρέπει λοιπόν να θέτουμε τα θέματα στις σωστές τους διαστάσεις όταν μιλούμε και αφιζητούμε την αποτελεσματικότητα της οδηγίας. Η οδηγία δεν προστατεύει τα υβριδικά είδη και όλο αυτό το θέμα μπορεί να επιληθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για το στατικό χαρακτήρα τώρα της οδηγίας και για το ότι υπάρχουν υπονοούμενα σύμφωνα με τα οποία η οδηγία είναι κατάλληλη και δεν μπορεί να ε, επιλύσει το πρόβλημα της βιοποικιλότητας. Εμείς έχουμε κάνει τις δικές μας αξιολογήσεις, θεωρούμε ότι οι οδηγίες αυτές ε, ταιριάζουν με τον προσδοκόμενο σκοπό, έχουμε ε, κάνει τα μαθήματά μας αν θέλετε και Ε, τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζουν την ε, ε, ίδια άποψη αλλά και του Συμβουλίου το οποίο Συμβουλίου έχει συμφωνήσει με αυτά τα συμπεράσματα. Άρα, να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτό το εργαλείο. Το ότι μπορεί να κυνηγάει κανείς κάποια είδη μόνο υπό το καθεστώς της παρέκκλησης, όπως είναι ο, ο κορμοράνος, και άλλα... Ε, το, ε, με το καθεστώς της παρέκκλησης δηλαδή μπορεί να το κυνηγάει, αυτό δεν είναι πρόβλημα από μόνο του και σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει επιπρόσθετο ε, διοικητικό ε, υπάρχουν δυνατότητες να ε, μειωθούν τα προβλήματα. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος μπορεί κανείς να προστατεύσει τις δραστηριότητες που υποφέρουν από τις καταστραφές του κορμοράνου, δηλαδή η το για παράδειγμα. Μπορεί να έχει προστατευτικά μέτρα για να αντισταθμίσει τις απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια, η χθιοκαλλιέργεια που προκαλεί η ανάδειξη των αποθεμάτων των κορμοράνων και η ενίσχυση αυτών. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές ρυθμίσεις και χειρισμοί που μπορούν να γίνουν. Πολύ έμφαση δίνεται στο σχέδιο ψηφίσματος για το μέλλον. είναι εγγενές χαρακτηριστικό του σχεδίου δράσης, δεν ασχολείται με θέματα κοινή γεωργικής πολιτικής. Οι δράσεις 9, 10 και 11 έχουν να κάνουν με την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλληλευτική πολιτική, πολιτική για τις περιφέρειες. Όλα αυτές οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί η χρηματοδότηση εκτείνεται μέχρι το 2020 και ως δαπάνη θα συνεχιστεί να δίδεται και μέχρι το 2022 και 2023. Άρα να προβληματιστούμε στο κατά πόσο θα βελτιώσουμε το πλαίσιο για το μέλλον. Έτσι όπως έχει το πλαίσιο χρηματοδότησης θα παραμείνει για τα επόμενα 5 και 6 χρόνια. Αυτό να το ξέρουμε. Άρα να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες για να ενισχύσουμε τη φύση και την βιοποικιλότητα. Και αυτός είναι και ο στόχος του σχεδίου δράση υπ' αυτή την έννοια. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις επεξηγήσεις σας. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 5η Σεπτεμβρίου στις 11. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 12 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στην δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Και περνάμε και στο τελευταίο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, πρόκειται για την εξέταση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. Εδώ επίσης έχουμε διάφορους συνεισήγητες και θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στο ΕΛΚΑ, στην κυρία Πιέτη Κάνεν, αλλά την αντικαθιστά κυρία Ντελέ, γιατί απουσιάζει κυρία Πιετικάνη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε, συνάδελφος Πιετικάινεν δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, ζητά συγγνώμη. Μου ζήτησε όμως να σας ενημερώσω εγώ για τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια περιβαλλοντική πολιτική και μάλιστα ισχυρή. Οπότε τα προβλήματα έγκυται στην εφαρμογή τη πολιτική αυτή και μάλιστα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έπρεπε υπέρ τη αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Εξού και η πρωτοβουλία αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και ε, δοκιμάζουμε, η οποία θα επιτρέψει την επίτευξη πολιτικών στόχων προκειμένου να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική νομοθεσία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες μέλη. Υπάρχουν όμως νέες εργασίες ε, για την ανάπτυξη της επισκόπησης αυτής, για την εφαρμογή της παραλωτικής πολιτικής. Οπότε περιμένουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, προκειμένου η επισκόπηση αυτή να γίνει πιο πλήρης, να καλύπτει και κάποια θέματα τα οποία λείπουν τώρα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι τα χημικά προϊόντα, οι βιομηχανικές εκπομπές, όλα αυτά να περιλαμβάνονται στην έκδοχη της επισκόπησης. Και αυτό για να διορθωθεί η κατάσταση. Όμως, επιπλέον πρέπει να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων. Στην πρόταση ψηφίσματος, λοιπόν, εμείς εντοπίζουμε τρία στοιχεία. Πρώτον, την αναγκαιότητα να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της περιοριστική πολιτικής θα πάει στην πολιτική ατζέντα. Δεύτερον, να ενισχυθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάει προς την ε, κατεύθυνση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και τρίτον να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων προκτικών και αξιολόγηση από τους ομοτήμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές. Η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνάδελφος νομίζω εξήγησε με πολύ σωστό τρόπο και θα μου επιτρέψει να είμαι σύντομη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι σοσιαλιστές και δημοκράτες εκτιμούν ιδιαιτέρως την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι στην Ευρώπη έχουμε κάποιες ρυθμίσεις για το περιβάλλον, ιδιαίτερα προχωρημένες και για την προστασία των πολιτών και για την προστασία των φυσικών μας πόρων. Όμως, πολύ συχνά δεν εφαρμόζεται πλήρως Και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα συγκρίνοντας τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Στα πλαίσια της εξέτασης εφαρμογής της νομοθεσίας υπάρχουν προβλήματα και στον τομέα των, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στον τομέα της ποιότητας του αέρα κτλ. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνδέσουμε και με την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει μια οδηγία για τα απόβλητα η οποία να γίνεται πραγματικά σεβαστή Η, εξέταση μας δείχνει λοιπόν ότι υπάρχουν ελλείψεις ανάλογα με τα διάφορα κράτη-μέλη και μας δίνει και κάποιες υποδείξεις έτσι ώστε οι ελλείψεις αυτές να καλυφθούν. Τα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά πολύ συχνά οφείλονται στην έλλειψη επενδύσεων και στα συστήματα διακυβέρνησης. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό να γίνει, αλλά έχει στρατηγική σημασία για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν η έκθεση αυτή να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα διάφορα κράτη-μέλη και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο εδώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για πολλές χώρες οι οποίες δεν σέβονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πολλές φορές οι χώρες αυτές δεν κάνουν αυτά τα οποία θα έπρεπε. Από την άλλη, καλό θα είναι να δούμε και η οδηγία αν έχει κάποια προβλήματα, ίσως να μην είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη σε προβλήματα στα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Τι ζητάμε λοιπόν, το είπε η συνάδελφος και το ξαναλέω και εγώ. Για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή, Ζητάμε πρώτον να διευρυθούν οι συγκεκριμένοι τομεί, τομείς ε, τους οποίους, ε, οι οποίοι μας απασχολούν και τους οποίους θέλουμε να καλύψουμε, ιδιαίτερα για την επίδραση ας πούμε χημικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να τις ανταλλάξουμε όπου αυτό είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε. Το ECR τώρα, ο κύριος Τσμάκερ. Ευχαριστώ. Υπόθηκε ήδη, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ισχυρή ε, περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά τα προβλήματα έγκυται στην εφαρμογή. Μιλήσαμε πριν για το δίκτυο Natura, για παράδειγμα. Αλλά η νομοθεσία που έχει να κάνει με τα απόβλητα, ε, τις εκπομπές και ένα σωρό άλλα παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε όπου η εφαρμογή δεν είναι ικανοποιητική. Συνεπώς, θα πρέπει να μιζάρουμε περισσότερο στην εφαρμογή. Αλλιώς όλοι αυτοί οι αυστηροί κανόνες και η καλή νομοθεσία πάει περίπατο. Είμαστε αυτό που λέμε στο Ολλανδικά χάρτινοι τίγρης. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η επισκόπηση εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο και να τη στηρίξουμε. Στο ψήφισμα υπάρχουν διάφορες προτάσεις για τη βελτίωση του μέσου αυτού. Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή, για παράδειγμα, να περιλάβει και την κλιματική πολιτική. Έπειτα, να υπάρξει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των δεδομένων. Επίσης, να υπάρχει πιο ενισχυμένη ανταλλαγή βέλτιστων προκτικών και αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων για να αποτελέσει πηγή έπνευσης και καινοτομίας. Είμαι σκιώδης για το πακέτο για τα απόβλητα και πάντα ε, πίστευα και εγώ ότι βέλτιστες πρακτικές και ανταλλαγή τους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να βοηθήσει πολλές κυβερνήσεις. Έχουμε να μάθουμε ένας από τον άλλον και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα. Η επισκόπηση εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει επίσης να είναι ένα μέσο που θα μπλέξει και το κοινό. Πρέπει και αυτό να ενημερώνεται. Η επιτυχία του βέβαια έχει να κάνει με την βούληση που διδειχθεί και με την εμπλοκή των διαφόρων πλευρών της περιφερειακής κυβέρνησης, της τοπικής κυβέρνησης που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά βέβαια το ζήτημα της εφαρμογής είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Γενικά όμως μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το ψήφισμα. Πιστεύω ότι δίνει ένα ισχυρό μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γερμπραντή, εκ μέρους των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι υπόθηκαν τα περισσότερα, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ πολλά. Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις για την αναγκαιότητα του νέου αυτού μέσου. Πιστεύω ότι είναι ε, μια πολύ έξυπνη κίνηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προσθέσει κάτι στην ε, νομοθετική εφαρμογή. Φοβάμαι ότι το τελευταίο μήνα τέλη Ιουλίου, όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε από την Πολωνία να σταματήσει ε, την υλοτομία, ο Πολωνός υπουργό είπε απλώ ότι δεν θα συμμορφωθεί. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ο περιφερειακός ε, νομικός ε, δρόμος είναι μεν αναγκαίο αλλά δεν είναι αποτελεσματικό. Οπότε βοηθάει η πρόταση αυτή, είναι μάλιστα αναγκαία, φοβάμαι. Χρειαζόμαστε όμω κάποια κριτήρια. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί και στην αρχική προσέγγιση χρειάζεται. Δηλαδή η βούληση των κρατών μελών. Το είπε και ο συνάδελφο τη Μακερ πριν από λίγο. Αν οι χώρε μέλη δεν είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με αυτό το μέσο ήπιας πολιτικής, ε, δεν θα είναι και αποτελεσματικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό, όχι μόνο προς την Επιτροπή, αλλά και προς τις χώρες μέλη. Είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν πλήρω με αυτή τη νέα προσέγγιση. Δεύτερον, έχει μεγάλη σημασία η διαφάνεια, γιατί Πολύ εύκολα μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από κλειστέ πόρτες με την επισκόπηση αυτή και τελικά να εξαρτώμεθα από εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πόσο αποτελεσματικό θα είναι το νέο μέσο. Η διαφάνεια όμως είναι ζωτικής σημασίας για μένα, γιατί έτσι και το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για την επιτυχία της νέας προσέγγισης. Αυτά. Και ελπίζω όντως να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο στο μέλλον. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει άλλος ε, συνεισηγητής παρόν, όμως έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Κάντεμπαχ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, να έχω μία παρατήρηση. Στο περιθώριο των όσων είπε ο κύριος μόλις τώρα, για τα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα έπρεπε να προωθήσουμε περισσότερο τους στόχους της νομοθεσίας αυτής. Γιατί υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Συχνά μιλώντας με τον κόσμο έχουμε την αίσθηση ότι η οικονομία, η βιομηχανία είναι το αντικείμενο στο οποίο δίνει περισσότερη έμφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το περιβάλλον. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές. Όχι για να ενοχλήσουμε την βιομηχανία, όχι για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις δικές μας προδιαγραφές, αλλά γιατί μακροπρόθεσμα υπάρχουν κάποιες καταστροφές που θα προκληθούν από τις εκπομπές αυτές. Δεν είναι για να ε, κερδίσουμε χρήματα από τη θεραπεία των ανθρώπων. Όχι, θέλουμε πρόληψη. Και πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, αν δεν υπάρχει τέτοια δράση περιβαλλοντική, ποιο θα είναι το κόστος, ποια θα είναι η ζημιά. Συχνά μιλάμε πόσο κοστίζει η κατάσταση ενός φίλτρου. Αλλά δεν μιλάμε για το κόστος των συνεπειών, άπαξ και δεν υπάρχει αυτό το φίλτρο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε ότι αν δεν δοθεί μία επένδυση μια συγκεκριμένη στιγμή, τελικά το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λέμε στον κόσμο και να υπάρχει πάντα στη συζήτηση που κάνουμε με το κοινό αυτή η σύνδεση. Και αυτό να το έχουμε υπόψη μας, όχι μόνο ενώπιση των επόμενων εκλογών, αλλά γενικά για να επιστήσουμε την προσοχή του κοινού. Πρόεδρος, υπάρχει κανένας άλλος που θέλει το λόγο. Α, παρακαλώ, η κύριε Ντάλη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα δύο σύντομες παρατηρήσεις να κάνουμε, έχοντας ακούσει τη συζήτηση και το διάλογο, μια παρατηρήση που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την αίσθηση ότι η επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ανακοίνωσή της για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν την περιβαλλοντική νομοθεσία είναι πολύ περιοριστική, δεν αναφέρεται ε, σε θέματα εκπομπών της βιομηχανίας, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τα σχετικά μέτρα, τα μέτρα για τη χημική βιομηχανία, για την κλιματική αλλαγή ε, για τη γεωργία, ε, την αλία, ε, την πολιτική για τις περιφέρειες. Δεν τα λαμβάνει υπόψη σε αυτά. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν πρέπει την περιβαλλοντική νομοθεσία να την εξετάσει σε τόσο στενό πλαίσιο, με, τόσο, με, με τέτοιες παραπίδες εντός εισαγωγικών θα έλεγα. Ε, χωρίς περίληψη άλλων τομέων. Έχουμε κανονισμούς και οδηγίες νομικώς δεσμευτικούς για το περιβαλλοντικό δίκαιο. Δυστυχώς όμως τα κράτη-μέλη τους αντιμετωπίζουν αυτός ως σαν να πρόκειται για απλές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι, είναι νομικώς δεσμευτικά κείμενα και ε, δεν υπονομεύει τίποτα περισσότερο την αξιοπιστία ενός δημόσιου φορέα από νομοθεσία που δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται. Μόνο έτσι χάνεται η αξιοπιστία ε, του φορέα, του οργανισμού ε, της Ευρώπης, του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόβλημα δηλαδή της συμμόρφωσης και των κανόνων που έθεσε ο Ευρωπαίος νομοθέτης υπάρχει διότι δεν τα τηρούν αυτά τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ακραδάντως ότι η συμμόρφωση και η εφαρμογή, αυτά είναι τα στοιχεία κλειδιά, αυτά είναι που πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά είναι αυτά στα οποία πρέπει να εστιάσουμε, έτσι ώστε για να έχουμε αποτελέσματα στην πραγματική μας ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προσωπικό συμφωνώ απολύτως με όλους τους προλαλήσαντες και με την ανάγκη επαιδαγωγικής και εκπαίδευσης ορισμένων και διδαχής τους. Ποιες κυρώσεις όμως θα εξετάσουμε. Πώς θα συνοδεύσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν δομικές δυσκολίες να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ίσως πρέπει να έχουμε τελικά περιβαλλοντική πολιτική κομμένη και ραμμένη στο χέρι γιατί είναι ε, λεπτοδουλιά, ε, βελονάκι αν θέλετε για να ταιριάζει ε, στις εκάστοτε δυσκολίες κάθε περιοχής. Ε, αν δεν υπάρχουν άλλοι βουλευτέ ε, που να θέλουν το λόγο, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο, στον Διευθυντή της ε, Αρμόδιας Διεύθυνσης. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, διότι μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εγκάρσια στήριξη. Όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν την πρωτοβουλία μας και θα μπορέσουν όλα αυτά τα θέματα να ψηφιστούν με ευρία πλειοψηφία μετά από τις προφορικές ερωτήσεις ε, και την απάντηση που έχει δοθεί σε αυτές. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μου επιτρέψετε να μιλήσω ε, στα αγγλικά για να διαβεβαιώσω τα μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τις καλύτερες προθέσεις και έχει τις καλύτερες προθέσεις όταν πρότεινε αυτή την πρωτοβουλία. Και πράγματι χρειαζόμαστε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, να τονίσουμε περισσότερο την εφαρμογή των εφιστάμενων περιβαλλοντικών κανόνων. Ήδη έχουμε αρκετούς κανόνες, ήδη έχουμε αρκετούς φιλόδοξους στόχους και είναι σημαντικό για να έχουμε αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών μας, αλλά και για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να έχουμε αξιοπιστία στα μάτια τρίτων χωρών, τα γεγονότα να συνάδουν με τα λόγια μας, οι πράξεις μας να ακολουθούν τα λόγια μας και να δείχνουμε ότι ακολουθούμε τις, και εκπληρώνουμε τις προσδοκίες των πολιτών και δρέπουν όλοι τα ωφέλη των περιβαλλοντικών κανόνων και θελήσαμε όλα αυτά να είναι και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την κατάλληλη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ε, αυξάνουμε την ε, ενσυναίσθηση, τη συνειδητοποίηση, τη γνώση. Ε, κατα, γίνεται ε, καλύτερα κατανοητός, κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι διάφοροι περιβαλλοντικοί κανόνες, οι οποίοι συχνά είναι πολύ περίπλοκοι γίνονται πιο εύληπτοι και πιο ευανάγνωστοι οι στόχοι των ε, περιβαλλοντικών κανόνων. Δεν θα πρέπει οι στόχοι ε, να ε, χάνουν σε ορατότητα, να μειώνεται η ορατότητά τους, να μην είναι εύληπτοι, ευανάγνωστοι και ευκόλως κατανοητοί και σε αυτό αποσκοπούμε με τις πολιτικές μας. Θέλουμε να ρίξουμε περισσότερο φως στον τρόπο με τον οποίο διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν οι κανόνες στους διάφορους τομείς. Περιβαλλοντική προστασία των υδάτων, πώς συνδέεται με την προστασία της φύσης, πώς συνδέεται με την περιβαλλοντική πολιτική. Πολλά μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, της δικής σας Επιτροπής, τόνισαν ότι υπάρχουν ε, σχέσεις άρρηκτες μεταξύ περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής για τη μεταφορά, για τις μεταφορές ή πολιτικής για τη γεωργία. Και όντως έτσι ισχύει. Ε, ε, υπάρχουν συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ περιβαλλοντικής πολιτικής και ε, πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Πολύ σημαντικές οι σχέσεις αυτές. Άρα να μην χάνουμε από, το, από μπροστά μας, από το μυαλό μας, το ευρύτερο πλαίσιο, τη συνολική εικόνα και να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Θελήσαμε επίσης να ρίξουμε φως στις κρυφές αιτίες πίσω από την κακή εφαρμογή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών κανόνων, που ενίοτε οι αιτίε είναι πολύ ευαίσθητες, είναι ένα λεπτό πολιτικό ζήτημα, ενίοτε υπάρχει τεράστια απώλεια πόρων ε, και απουσία πόρων και δυναμία εφαρμογής αυτών δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να αποφασίσει ποιος θα έχει αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία γιατί οι εθνικές αρχές πρέπει να αυτό να το πράττουν. Όταν όμως δίδεται εξουσία και αρμοδιότητα στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση τότε αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από κατάλληλους πόρους οικονομικούς και εργαλεία για να μπορέσει να εφαρμοστεί η ε, νομοθεσία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη την ευθύνη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας έχουν την ευθύνη αυτή οι περιφέρειες και οι δήμοι. Τα ίδια τα κράτη-μέλη σε κεντρικό επίπεδο πολύ συχνά έχουν μόνο ε, κρατήσει για τον εαυτό τους το δικαίωμα της εποπτείας Άρα θα πρέπει οι περιφέρειες και οι δήμοι να έχουν τα απαραίτητα κονδύλια, αλλά και την ικανότητα, τους ανθρώπινους πόρους με τεχνογνωσία ε, και προσόντα για να μπορούν να την εφαρμόσουν αυτή την περιβαλλοντική νομοθεσία. Αυτά θέλουμε να το τονίσουμε. Και βεβαίως υπάρχουν ευθύνες για την επιβολή του νόμου, ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις συνθήκες ε, έχουμε τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Και ορισμένοι εταίροι μας από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις φοβούνταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει πιο μαλακή με αυτές τις προτάσεις και δεν θα κοιτάζει να επιβάλλει τον νόμο με αυστηρότητα. Όχι. Εμείς θελήσαμε να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να ενημερώσουμε όλους, να αφυπνίσουμε όλους η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας χρειάζεται χρόνια για να γίνει. Δεν αρκεί να αλλάξουμε τους κανόνες. Πολύ συχνά πρέπει να γίνουν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές για τα αστικά λίματα, για τη διαχείριση των υδάτιτων πόρων, για τις μεταφορές, για τη ρήμανση την ατμοσφαιρική και άλλη από τη συγκοινωνία της μεταφορές, για τη διαχείριση αποβλήτων. Πολλές φορές για να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική νομοθεσία οι επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν παίρνουν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν. Γι' αυτό έχουμε το σύστημα κύριε προειδοποίησης για να προλάβουμε καταστάσεις, όχι για να μειώσουμε την αρμοδιότητα και εξουσία μας την, ως, προς, την επιβολή της νομοθεσίας. Από εκεί και πέρα, διαβεβαιώνω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν σήμερα το λόγο ότι το μήνυμα ελήφθη και ε, θα έχουμε μια δεύτερη έκδοση της έκθεσης αυτής όπου θα αναφέρουμε τα προσκόμματα, τα εμπόδια, τις ελλείψεις, τα κενά. Η πρώτη αυτή έκθεση ήταν και δοκιμαστική, να δούμε κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα και τις δυνάμεις να διαχειριστούμε την συνολική εικόνα, το άθροισμα των δεδομένων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους τομείς, μεταφορές ε, και λοιπά ενέργεια να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα με τα κράτη-μέλη. Ακούμε το μήνυμά σας, το λαμβάνουμε, το σημειώνουμε. Χρειάζεται συγκρισιμότητα των δεδομένων στις εκθέσεις αναχώρα. Βλέπετε στατιστικές που διατρέχουν ολόκληρη τη χώρα είναι αναχώρες. Όχι σε όλους τους τομείς, αλλά υπάρχουν να σας εφιστήσω την προσοχή σε εσάς τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν πρόκειται περί διαγωνισμού ομορφιάς εδώ. Δεν πρόκειται περί αγώνα δρόμου κούρσας για την πρωτιά μεταξύ των κρατών μελών. Όχι. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή ε, στο πού βρίσκεται η χή χώρα στο πλαίσιο το ευρύτερο των υπολείπων χωρών, αν είναι στο α, στο β, το γ. Δεν θέλουμε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, αλλά να κάνουμε πιο ουσιαστική ανάλυση σε βάθος. Και συμφωνούμε, πρέπει να γίνει ανταλλαγή των καλών πρακτικών. Όσοι έχουν δει τη συνοπτική σελίδα στην αρχή της έκθεσης αναχώρα ε, θα διαβάσετε ότι δύο-τρεις παραγράφους τις έχουμε αφιερώσει στα στο να πούμε σε ποια σημεία η χώρα είχε και την καλύτερη επίδοση. Συνοψίζουμε δηλαδή τα περισσότερα, βασικά επιτεύγματα, αλλά και τα βασικά εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδι για την κάθε χώρα. Συμφωνούμε για τις βέλτιστες πρακτικές και έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο, την ανταλλαγή μεταξύ ομολόγων, -peer exchange και θεωρούμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο θα ενεργοποιηθεί η χρήση αυτού του εργαλείου ε, μεταξύ ομολόγων. Θετικός ήταν ο αντίκτυπος από το Συμβούλιο. Τα λόγια μας βρήκαν απήχηση στο Συμβούλιο και είχαμε ήδη διάφορες διμερείς συναντήσεις με διάφορες χώρες, με διάφορα κράτη-μέλη και θα συνεχίσουμε να ε, συσκεπτόμεθα ε, διμερώς ε, κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου του 17 και της άνοιξης του 18. Όταν εξετάζει κανείς το διμερή διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκάστοτε κράτους μέλους, πρέπει να απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα της χώρας, όχι μόνο στις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρέπει να μιλήσει και στον Υπουργό Οικοτομίας, στον Υπουργό Γεωργίας, στον Υπουργό Μεταφορών και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να μην μιλήσει μόνο ε, στις περιβαλλοντικές αλλά και στις οργανώσεις των εργοδοτών, των βιομηχανιών, των κλάδων, των οικονομικών φορέων να εμπλακούν πολλές και διαφορετικές δηλαδή εθνικές αρχές από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπρόσωποι από ε, όλους αυτούς τους φορείς για να ε, ξεπεράσουμε τα στενά όρια της περιβαλλοντικής κοινότητας και να βρούμε περισσότερη απήχηση στα λόγια μας. Στο Βέλγιο ήταν πολύ θετική η εμπειρία μας, στην Ουγγαρία επίσης πολύ θετική η εμπειρία μας, ε, η Τσεχία, η Δημοκρατία της Τσεχίας επίσης, προετοιμαζόμαστε και ετοιμαζόμαστε για πιο θετικούς και ανοιχτούς επικοδομητικούς δημιουργικούς διαλόγους με το Λουξεμβούργο και με τη Φιλανδία αυτή τη στιγμή που θα ξεπεράσουν τα στενά όρια της περιβαλλοντικής κοινότητας. Δεν θέλουμε μόνο η περιβαλλοντική κοινότητα σε κάθε χώρα να είναι ο συνομιλητής μας. Και θα ήθελα να σας απαντήσω κυρία Πρόεδρε στη δική σας ερώτηση για τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι αυτές που έχουν προσδιοριστεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση παράβασης ε, των κανόνων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να ασκήσει το δικαίωμά της για τη διαδικασία επιπαραβάση ε, όταν εντοπίζει προβλήματα ε, κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και λαμβάνουμε υπόψη τα ευρήματα στα οποία έχουμε καταλήξει στην εξέταση και αναθεώρηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να σας πω ότι έχουμε ήδη ε, δημιουργήσει αυτό το εργαλείο ε, αρρωγής μεταξύ ομολόγων, peer-to-peer -peer assistance και exchange. Θα το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά και θεωρούμε ότι θα φέρει καρπούς. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξή της κατά την, ε, κατά την ε, επανεξέταση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα σας είμαστε ευγνώμων εάν στηρίξετε τη δουλειά μας για την εφαρμογή. Ε, θέλουμε να συμπεριλάβετε στην πολιτική σας ατζέντα, στην εκλογική σας περιφέρεια, τη στήριξη για την αταλάντευτη και σταθερά προσιλωμένη εφαρμογή, αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε ε, ως προς τούτο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς για τις λεπτομερείς εξηγήσεις που μας δώσατε. Οπότε σας υπενθυμίζω τις ημερομηνίε τώρα όσον αφορά την πρόταση αυτή ψηφίσματος. Πρώτα απ' όλα, η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου στις 11. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 11 ή 12 Οκτωβρίου και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν υπάρχουν διάφορα, οπότε Ολοκληρώνουμε εδώ την συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ τους βουλευτές που παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής. Και σας υπενθυμίζω ότι θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Ως ήθιστε. Ευχαριστώ. Merci.